αύριο στις 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητάω την κατανόησή σας για το ότι για τεχνικούς λόγους θα διακόψουμε για δύο λεπτά και θα επαναλάβουμε αμέσως. Δύο λεπτάκια. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σα ευχαριστώ για την υπομονή σα. Το τεχνικό ζήτημα αντιμετωπίστηκε. Συνεχίζουμε. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Κοινή συζήτηση για τι διμερεί ρήτρε διασφάλιση και μηχανισμοί σταθεροποίηση για τι μπανάνε. Θα συζητήσουμε τι εκθέσει Λάγκε για τις εφαρμογές ε, των διμερών συμφωνιών μεταξύ της Κολομβίας και του Περού και της ε, Κεντρικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ο κύριος Λάγκη για 4 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι σας ευχαριστώ για το ότι είστε εδώ πέρα απόψε και μπορούμε να συζητήσουμε κάτι το οποίο προφανώς ε, δεν απασχολεί και ιδιαίτερα την Ολομέλεια. Ασχολούμαστε με τις ρήτρες διασφάλισης και μηχανισμούς σταθεροποίησης σε ζητήματα δηλαδή τα οποία αναφέρονται στη συνθήκη της Λισαβόνας αλλά εξακολουθεί να μην είναι ξεκάθαρο το ποιο θεσμικό όργανο έχει πια αρμοδιότητα και τι ρυθμίζεται που έτσι έχουμε παραδείγματο χάρη νομοθεσία μέσω της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας και κάποια σημεία ενσωματώνονται θέματα δηλαδή τα οποία είχαν ενσωματωθεί ε, μετά από μια απόφαση Συμβουλίου λάθος στην συνθήκη. Οπότε νομίζω πως είναι καλή άσκηση συνολικά να δούμε τις ρήτρε διασφάλισης για τις συμφωνίες με Κολομβία και Περού. Γιατί αφενός βεβαίως απέναντι στην Κολομβία και στο Περού θέτουμε απαιτήσει σε αυτές τις χώρες και πρέπει να δούμε πώς θα εκπληρώσουμε λογικά και τις απαιτήσεις που θέτουμε στους αυτούς μας. Και θεωρώ σημαντικό είναι να παραμείνει η ρήτρα διασφάλισης και πρακτική να εφαρμόζεται. Δεν είναι να γράφουμε πράγματα που δεν θα ισχύσουν ποτέ γιατί έτσι είχε γίνει στο παρελθόν. Γι' αυτό αυτό το οποίο έχουμε εμείς ως δυνατότητα διαμόρφωση πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε οι ρήτα διασφάλιση και οι μηχανισμοί σταθεροποίησης να βγουν από την σκόνη των φοριαμών και να αποκτήσουν μια πραγματική ζωή. Και εδώ πέρα έχουμε λοιπόν πέντε σημεία κύριε Επίτροπε. Πρώτον, να δούμε ποια είναι τα κριτήρια για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ασφαλείας. Είμαι δε τα πεπισμένος πως όταν διαπιστώνουμε πως υπάρχει εμπειριασμός της αγοράς θα πρέπει να δούμε και το ζήτημα των κοινωνικών προδιαγραφών γιατί βεβαίως αν δεν υπάρχουν και κάποιοι κοινωνικοί όροι υπάρχει κάποιο dumping και κάποιο άδικο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και άρα ε, ισχύει αυτομάτως η ρήτρα διασφάλισης. Δεύτερον, αν είναι να εφαρμοστεί η Λισαβόνα πρέπει να δούμε και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι σαφές πως εμείς όπως και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, επιζητούμε το δικαίωμα να μπορούμε να ξεκινήσουμε μια έρευνα. Τρίτον, αν μιλάμε σοβαρά περί διαφάνειας, νομίζω πως πρέπει να δούμε και το πώς θα συμπεριληφθεί και η κοινωνία των πολιτών σε έναν διάλογο για να εξετάσει και την συμφωνία παραδείγματο χάρη με την Κολομβία και το Περού. Και θέλουμε άρα να ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Κύριε Επίτροπε, εσεί παραπέμπετε πάντα στο μοντέλο της ρήτρα διασφάλισης με την Κορέα. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε κάποια παρακολούθηση και εκθέσεις. Ε, το άρθρο 11 λοιπόν της συμφωνίας με την Κορέα το έχετε ξεχάσει. Εμείς θα θέλαμε να διασφαλιστεί εδώ πέρα. Και πέμπτον έχουμε την διασφάλιση των παραγωγών μπανάνας στις ευρωπαϊκές ε, περιφέρειες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Κατόπιν ο κύριος Λάχιθρη για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κεντρική, στην Κεντρική Αμερική η κατάσταση είναι παρόμοια με το Περού και την Κολομβία και άρα αυτά τα οποία ανέφερε ο συνάδελφος ισχύουν και για τη δική μου έκθεση και άρα θα είμαι κάπως συντομότερος θεωρώ πως η όλη συζήτηση έχει δύο πτυχές. Μια τεχνική και μια άλλη πτυχή, η οποία είναι πολύ ευρύτερη. Η τεχνική πτυχή είναι σχετικά απλή. Η ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να διασφαλίζει τους Ευρωπαίους παραγωγούς με το άνοιγμα της αγοράς από τον άδικο και αθέμητο ανταγωνισμό. Διατυπώσαμε λοιπόν τη ρήτρα διασφάλιση κατά τρόπο ώστε να λειτουργεί, αλλά και βεβαίω ε, με τρόπο ώστε να λειτουργεί και το ελεύθερο εμπόριο. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά νομίζω πως καταλήξαμε σε καλούς συμβιβασμούς για να βρούμε μια λύση. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη πτυχή, μια φιλοσοφική θα έλεγα, που είναι όμως και αυτή. Το θέμα δηλαδή αρχής, το οποίο είναι η εμπορική πολιτική πρέπει να είναι μόνο εμπορική ή να είναι κάτι περισσότερο. Αυτό το ερώτημα μας απασχόλησε και σε αυτή τη συζήτηση για τις ρήτρες διασφάλισης και πρέπει βεβαίως να παρατηρήσω πως οι ρήτρες διασφάλισης είναι ένα μικρό τμήμα αυτής της συνολικής συμφωνίας με την Κεντρική Αμερική. Και αυτό ήταν ο λόγο για τον οποίο είπαμε όχι, ακόμα και η ρήτρα διασφάλιση πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από μια ρήτρα διασφάλιση. Πρέπει να προσπαθεί να επηρεάζει πράγματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, την οικολογική πτυχή. Υπάρχουν κάποιοι νομικοί οι οποίοι λένε «Μα τι δουλειά έχουν αυτά σε μια ρήτρα διασφάλισης». Έχουν δουλειά όμως. Γιατί, γιατί μια τέτοια ρήτρα τελικά, το ανέφερε και ο κύριος Λάγκε, έχει στόχο να προστατεύσει θέσεις εργασίας Ευρωπαίων. Και για να γίνει αυτό πρέπει να φροντίσουμε να βελτιωθούν αυτά τα πράγματα, οι κοινωνικές συνθήκες, τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες εταίρους μας. Το μεγάλο ερώτημα είναι βεβαίως και εδώ πέρα κάποιοι συνάδελφοι διαφωνούν, σε ποιο βαθμό οι προσπάθειες αυτές επηρεασμού άλλων χωρών μέσω της εμπορικής πολιτικής θα μπορούν να φτάσουν. Δεν μπορούμε μέσω της εμπορικής πολιτικής να ασχολούμαστε με ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής άλλων χωρών. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα προς μία σωστή κατεύθυνση. Αυτό προσπαθήσαμε. Υπάρχουν βεβαίως διαφορετικές κατευθύνσεις. Ε, αυτό το οποίο προέκυψε είναι ένας συμβιβασμός, νομίζω λογικός και γι' αυτό θεωρώ πως λογικό θα ήταν να υπερψηφίσουμε αύριο ε, αυτές τις ρήτρες διασφάλισης. Η δε συζήτηση για το οριστικό αποτέλεσμα θα είναι οπωσδήποτε πιο έντονη. Στις ρήτρες διασφάλισης όμως νομίζω πως πρέπει να δούμε πως είναι απλά οι ρήτρες διασφάλισης και όχι η συνολική συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Επιτροπός, ο κύριος Δικούχτη έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τον κύριο Λάγκη και τον κύριο Λάιχτφιντ για τη δουλειά που έκαναν για αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δίνετε για να διευκρινίσουμε τα ε, κρεμή θέματα για την ε, υιοθέτηση των ε, κανονισμών για τις διμερείς ρήτρες διασφάλισης με το Περού, την Κολομβία και την Κεντρική Αμερική. Το Ιούνιο υπογράφτηκαν και αμέσως το Κοινοβούλιο αποφάθηκε μέσω μιας διαδικασίας συνένεσης. Πριν εξηγήσω τη σημασία το, τη υιοθέτηση αυτών των κανονισμών διασφάλισης θα ήθελα ακόμα να σα τονίσω ότι έχουν μεγάλη σημασία αυτοί οι κανονισμοί για αυτέ τι δύο περιοχέ της Λατινική Αμερική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμφωνία με την ε, Κεντρική Αμερική και το Περού και την Κολομβία έχουν αναβαθμίσει τι σχέσει μεταξύ ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των δύο αυτών περιοχών. Εμπορικό πώ αυτέ οι συμφωνίε θέλουν να ανοίξουν τι ε, αγορέ για αγαθά υπηρεσίε, κρατικέ προμήθειε και επενδύσει. Ε, μιλάμε για ε, γεωργικά προϊόντα, αλληλευτικά προϊόντα που και τα γεωργικά προϊόντα θα προωθηθούν γιατί θα κάνουμε μεγάλες ε, παραχωρήσεις σε ποσοστώσεις. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε εμπορικούς κανόνες που είναι πολύ προβλέψιμοι Αυτές οι συμφωνίες θα μας ε, παρέχουν ένα πλαίσιο προβλέψιμο, ε, μια δέσμη εμπορικών κανόνων μέσα στους οποίους οι εμπορικοί παράγοντες, ε, οι ενδιαφερόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις χώρες αυτές μπορούν να υποφεληθούν. Οι καθαρές εμπορικές ροές θα ξεπεράσουν τα εμπορικά όρια, γιατί θα εξασφαλίσουν και την υφοροανάπτυξη ε, και θα έχουν και ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να μπω τώρα στο θέμα της υιοθέτηση των ε, διμερών ε, κανονισμών διασφάλισης. Ο στόχος αυτού του κανονισμού είναι να έχουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για τη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης των δασμών έχουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα λόγω των εισαγωγών για να εφαρμόσουμε αυτές τις διατάξεις, χρειαζόμαστε τους καονισμούς μάλλον. Ε, καλωσορίσουμε τις αρχές που αναφέρουν οι συγητές όταν, ότι θα πρέπει δηλαδή μέσω τροπολογιών να προσκολήσουμε περισσότερο ε, στο μοντέλο της Κορέας, αλλά να λάβουμε υπόψη μας και τις ιδιαιτερότητες αυτών των περιοχών. Οι εφαρμοστικοί κανονισμοί επίσης δεν μπορούν να έρχονται σε αντίφαση με τις συμφωνίες και με τους τις δεσμεύσεις και τους κανόνες του ΠΟΕ. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι η κοινοβουλευτική αυτή συζήτηση για αυτούς τους κανονισμούς είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν θα πρέπει όμως ε, να είναι η ευκαιρία για να ξανανοίξουν ερωτήσεις που έχουν ρυθμιστεί όπως σεβασμός των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Όπως ξέρετε τα θέματα αυτά καλύπτονται ήδη από τις συμφωνίες. Ε, στο ψήφισμα του Ιουνίου του 2012 επίσης το Κοινοβούλιο εξέφρασε την πολιτική γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε για, το, και εμείς αλλά και οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις των δύο χωρών του Περού και της ε, Κολομβίας. Εμείς έχουμε λάβει υπόψη μας αυτό το ψήφισμα και συνεργαζόμαστε με τις δύο χώρες για να εφαρμοστεί. Για να ολοκληρώσω, θέλω να σα εκφράσω την ευχή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κομισιόν, το Συμβούλιο θα έχουν μια καλή συνεργασία στα πλαίσια του μερού διαλόγου που θα ξεκινήσει σύντομα, ούτω ώστε όλε αυτέ οι προποθέσει ε, να υπάρχουν, ε, ούτω ώστε να συνενέσει και το Κοινοβούλιο με αυτέ τι συμφωνίε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Κατόπιν για την Επιτροπή Γεωργίας, ο κύριος Άντροβερ. Ευχαριστώ πολύ ξεκινώντας από τη βάση πως οι συμφωνίες αυτές με την Κεντρική Αμερική, το Περό και την Κολομβία είναι εξαιρετικά βλαβερές για τους Ευρωπαίους παραγωγούς μπανάνας και κυρίως για τα Κανάρια νησιά, που βρίσκονται εκτός της εξισωτικής ε, αποζημίωσης ΠΟΣΕΗ που ελπίζω θα τους χορηγηθεί αργότερα. Παρόλα αυτά θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί πολλές από τις προτάσεις μας συμπεριλέφθηκαν εδώ. Άρα λοιπόν οι ρήτρες διασφάλισης έχουν βελτιωθεί και έχουμε και το μηχανισμό σταθεροποίησης. Μεγαλύτερη διαφάνεια και μια εξαντλητική παρακολούθηση των εισαγωγών μπανάνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποια προληπτικά μέτρα επιτήρησης που θα εφαρμόζονται. Έχουμε λοιπόν και την ειτήσια έκθεση για τη ρήτρα που θα πρέπει κατά τη γνώμη να συμπεριλαμβάνει και μία παρακολούθηση το πώς οι εισαγωγές μπανάνας επηρεάζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή. Όλα αυτά επαναλαμβάνουν είναι σημαντικά. Η παραγωγή της Ευρώπης που είναι από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές αυτή τη στιγμή αυτή τη δύσκολη στιγμή χρειάζεται τη βοήθειά μας. Πολύ δρόμο έχω έχουμε ακόμα να κάνουμε, αλλά το βήμα το οποίο σημειώσαμε ήταν εξαιρετικά σημαντικό. ευχαριστώ. Για το ΕΛΚ τον λόγο έχει ο κύριος Ζάλβα Βιντεγκάιν. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η προβλεπόμενη έγκριση των τροπολογιών ε, για τα κείμενα αυτή για τα μπενάνα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός στα πλαίσια της προσπάθειας έγκρισης από το Κοινοβουλίο των Συμφωνιών με την Κεντρική Αμερική, την Κολομβία και το Περού, που είναι συμφωνίες σκληριά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με τα εμπρόδο που έχει κάνει η Κολομβία, γιατί αυτό φαίνεται και από την ανακοίνωση που εγκρίναμε στις 13 Ιουνίου ε, και μαζί με τη στήριξη που προσέφεραν ε, και το Περού και οι χώρες Κεντρικής Αμερικής ε, σε αυτόν τον κανονισμό θα πρέπει να μας οδηγήσουν στην πλήρη έγκριση και η υπογραφή αυτών των συμφωνιών. Επιτρέπουν αυτές οι ρήτρε τους παραγωγούς μας να προσαρμοστούν σταδιακά σε μια ελεύθερη εμπορία των προϊόντων αυτών που θα μας ευνοήσει όλους. Αυτή τη στιγμή οι ασιατικές χώρες και η ΙΠΑ ε, ε, υπογράφουν συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τις ε, ε, χώρες Κεντρικής Αμερικής. Ε, και επίσης υπογράφουν η Κολομβία και το Περού ελεύθερη εμπορία αυτών των προϊόντων με τη ΣΥΠΑ. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούμε, δεν επιτρέπεται εμείς να συνεχίσουμε να χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Και γι' αυτό βεβαίως κατανοώ τις ανησυχίες βέβαια του κλάδου στην Ευρώπη, αλλά πιστεύω ότι η είσοδος αυτών των συμφωνιών θα μας ευνοήσει, επαναλαμβάνω όλους. Ευχαριστώ για τους σοσιαλδημοκράτες. Για ένα λεπτό τον ο κύριος Σούστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Λίχτριτ. Η διαπραγμάτευση της εμπορικής συμφωνίας με την Κολομβία και το Περού και με την Κεντρική Αμερική και οι μηχανισμοί σταθεροποίησης, οι ρήτρε διασφάλισης ε, μας κράτησαν έτσι σε αναταραχή πολλούς από εμά που ανέχουμε και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ. Νομίζω ότι υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε διάφορες ανάγκες. Καταρχάς, ε, ελεύθερο εμπόριο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 προστασία του κοινοτικού συμφέροντος, ε, πρόθεση του διεθνού εμπορίου, τόσο ώστε να υπάρχει μια ανάπτυξη που να βασίζεται στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδίω αυτοί οι κανονισμοί έχουν σαν σκοπό να προστατεύσουν τι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ακόμα δηλαδή επομένω και του ε, εργαζομένου, του ε, γεωργού μα, ειδικά των πιο περιφερειακών περιοχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι μηχανισμοί σταθεροποίηση και διασφάλιση, παρότι έχουν χρονικό περιορισμό, πιστεύω ότι ο χρονικός αυτός ορίζοντα επαρκεί ώστε να προσαρμοστούμε στην προκλεπόμενη απελευθέρωση. Στο μεταξύ, να βοηθήσουμε και τη σημαντική ανάπτυξη, των εξαγωγών ε, των διαφερμένων χωρών. Γι' αυτό λοιπόν ε, σας δίνουμε την θετική μας γνώμη και υπερψηφίζουμε τις εκθέσεις αυτές. Σας ευχαριστώ για την άλλη... για ένα μισή λεπτό. Κυρία Πίτερ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πότε είναι ένα καυτό θέμα, όχι και τόσο καυτό, όταν μιλάμε για τι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες των Άνδεων, για μία φορά το καυτό θέμα δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά οι μπανάνε. Όπω με όλε τις εμπορικές συμφωνίες πρέπει να διασφαλίσουμε πω με το άνοιγμα των αγορών μα επιτρέπουμε στι ευρωπαϊκέ εταιρείε και πραγωγού χρόνο προσαρμογή. Καλωσορίζω λοιπόν τις ε, ρήτρες διασφάλισης ε, στις συμφωνίες με την Κολομβία, το Περού και την Κεντρική Αμερική. Όμως είχαμε πικρή εμπειρία από τους πολέμους της μπανάνας, οπότε θα πρέπει να μην πατήσουμε ξανά την μπανανόφλουδα. Η ομάδα μου, οι φιλελεύθεροι και οι δημοκράτες θα καταψηφίσουν τις ε, τροπολογίες οι οποίες ε, κάνουν τα όρια αυτόματες ποσοστώσεις πρέπει να δώσουμε στην Κομισιόν την ευελιξία να αποφασίζει εάν παραδείγματο χάρη μια πλημμυρίδα εισαγωγών από την Κωνσταντίνα ή άλλη χώρα βλάπτει του Ευρωπαίου παραγωγού ή απλά αντισταθμίζει τη μειωμένη παραγωγή σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει πω πρέπει να δώσουμε ε, λευκό εξοδότηση στην Κομισιόν. Μάλιστα υποστηρίζω τι τροπολογίε που δίνουν μεγαλύτερο λόγο στην κοινωνία των πολιτών και στο Κοινοβούλιο έτσι ώστε να παρακολουθούμε την Κομισιόν και οι φωνέ των απλών πολιτών να γίνονται σεβαστές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη ομιλήτρια για τους ε, πράσινους, η κυρία Κέλλερ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και στην Κεντρική Αμερική και στο Περού και στην Κολομβία υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμείς ως ευρωβουλευτές δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας. Το ότι ξέφυγαν από τον ευρωπαϊκό οδικό χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα Κολομβία και το Περού είναι κάτι το αρνητικό και πρέπει να έχει αποτελέσματα και να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα του θα χάρη την καταδίκη των εγκληματιών και βεβαίως πριν από την ψηφοφορία πρέπει να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Επίσης θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό πως υπάρχουν εδώ πέρα περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές και όχι μόνο περιορισμούς τόνων για τις μπανάνες. Αλλά αυτά πρέπει να επιβεβαιωθούν και στον τριμερή διάλογο, αλλιώς δεν έχουν καμία αξία. Πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα για να βελτιώσει την κατάσταση επιτόπου για το πληθυσμό εκεί πέρα. Γι' αυτό πριν από κάθε διαπραγμάτευση θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση αντικτύπου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και του αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία συνάδελφε για την ΚΟΕ για 1,5 λεπτό. Τον λόγο έχει ο κύριος Ομαρζή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Δεν είμαι εξίσου αισιόδοξο με όσου πιστεύουν πω αυτέ οι ρήτρε ασφάλιση με τον τρόπο που έχουν τροποποιηθεί είναι επαρκεί για να προστατεύσουν την κοινοτική παραγωγή μπανάνα. Μόνο το όνομα φέρουν από τη διασφάλιση. Δεν διασφαλίζουν γιατί με τις συμφωνίες αυτές δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός ούτε των υπογραφών ε, την ε, συμφωνία ούτε της Κομισιόν. Ξέρετε με ποιο τρόπο θα πλήξουν τις μπανάνες από τις απομακρυσμένες μας περιοχές και τις υπερπόντιες περιοχές αυτές οι συμφωνίες είναι πλέον ε, σχεδόν εικονική η παραγωγή. Ε, δεν νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να χειροκροτήσουμε το γεγονός πως αυτή τη στιγμή προσφέρουμε κάποια προσπάθεια στήριξης. Να σας πω πως υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός από τις χώρες εξαγωγής μπανάνας από την Λατινική Αμερική και αυτή η τυφλή απελευθέρωση των συναλλαγών που προσπαθεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας εξυπηρετεί καθόλου. Σας υπενθυμίζω ότι έχω καταθέσει τροπολογίες έτσι ώστε να προστατεύσουμε κατά το ελάχιστο και τις θέσεις εργασίας στις περιοχές παραγωγής μπανάνας στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια αλλά και την παραγωγή την ίδια. Κύριε συνάδελφε, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Λάχιστριτ. Ε, κύριε Λάχιστριτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, παίρνω σας σοβαρά αυτά τα οποία λέτε αν και εγώ πάντα προσπαθώ να καταφέρω το καλύτερο, ειδικά όταν μιλάμε για κοινωνικές συνθήκες, προστασία των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, αλλά και στις χώρες εταίρους. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία που έπρεπε να πετύχουμε παραπάνω για να μπορέσετε εσείς να συμφωνήσετε με αυτές τις ρήτρε διασφάλισης. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας κατέφθεται κάποιε τροπολογίε ακριβώ για αυτό το λόγο, οι οποίε δεν ε, υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή ΙΝΤΑ και θα ψηφιστούν αύριο. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την δρομολόγηση των ρητρών διασφάλιση. Υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο που αφήνουμε προς εκτίμηση. Αυτή είναι και η άποψή μου και πιστεύουν και κάποια άλλα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πιστεύουν επίσης και οι επαγγελματίες της μπανάνας ότι το περιθώριο αυτό είναι πολύ μεγάλο. Για την τρομολόγηση αυτών των ρητρών διασφάλιση, καλό θα ήταν να είχαμε βάλει κριτήρια λίγο πιο περιοριστικά. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο, έσβησε το μικρόφωνο προ το παρόν του, του ομιλητή. Δεν το ακούσαμε το δεύτερο στοιχείο γιατί έσβησε το μικρόφωνο. Καλώ. Κατόπιν για ένα λεπτό τον λόγο έχει η κυρία Αντρέ Μπαρέα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η εμπορική συμφωνία με την Κολομβία, Περού και την Κεντρική Αμερική είναι σημαντική και οι ρήτρε διασφάλιση, αυτό που προσπαθούν να κάνουν με τι τροπολογίε που καταθέσαμε, είναι να είναι ευέλικτη, να είναι εύκολη και να προσφέρει κάποιε εγγυήσει. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή σύμφωνα με τις συνθήκες και να δημιουργήσουμε κάποιους μηχανισμούς εξασφάλισης για την ευρωπαϊκή παραγωγή αλλά και για την παραγωγή μπανάνας στις χώρες με τις οποίες υπογράψαμε τη συμφωνία. Είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τις υπερπόντιες περιοχές γιατί δεν έχουμε εκεί διαφοροποιημένες καλλιέργειες, γιατί είναι πολύ σημαντικές ε, οι καλλιέργειες αυτές για πάνω από 10.000 άμεσες θέσεις εργασίας και 35.000 έμεσες στην Ισπανία, σε μια περιοχή που πλήττεται πάρα πολύ από την ανεργία και που έχει κάποια ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Δηλαδή η μπανάνα από τα Κανάρια ε, είναι πολύ ιδιαίτερη και σε επίπεδο καλλιέργειας και σε επίπεδο γεύση, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ε, τη χρησιμοποιούμε στη γαστρονομία. Να υπογράψουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία το εμπόριο είναι σημαντικό για την ανάπτυξη και η ανάπτυξη την εργασιακά, δικαιώματα, βιωσιμότητα και βεβαίως το κέρδος να επιστρέψει στον παραγωγό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Τυρολιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συζητητές για τη δουλειά που έκαναν για αυτό το θέμα χρειαζόταν ε, με βάση την πρόταση της Κομισιόν. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στις υπερπόντιες περιοχές που πλήττονται από τον ανταγωνισμό των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα στο κοινοβούλιο μας να συζητήσουμε για τη ρήτρα διασφάλισης, για τους τρόπους ομολόγησή της. Δεν μιλάμε για τα κοινωνικά θέματα, για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η αυριανή ψήφος να επικυρώσει α, τα θετικά στοιχεία που έχει πει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, η ΙΝΤΑ. Ε, όμως δεν αρκούν αυτά, γιατί τα κατόφλια δρομολόγησης των δύο κανονισμών είναι τόσο ψηλά που καθιστούν, αυτού αυτούς τους μηχανισμούς διασφάλισης σχεδόν ανεφάρμοστους. Επίσης, η Κομισιόν θα πρέπει να προβλέψει ένα επιπλέον χρηματοδοτικό ποσό, ούτως ώστε να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα το, της κοινοτικής μπανάνας. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλές της απασχόληση υπάρχουν σε αυτές τις ευρωπαϊκές περιοχές, ε, που μην ξεχνάτε ότι πλήττονται από μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Ευχαριστώ. Danke, σας ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, τώρα δεν θέλω να ξύνομαι στην ε, γκλίτσα του Τσοπάνη, αλλά νομίζω πως κανείς δεν έχει ζητήσει το λόγο στο KHDI. Οπότε θα δώσω τον λόγο στον ε, κύριο Επίτροπο. Παρακαλώ. Thank you, President. Uh, first of all, let me... Θα ήθελα καταρχήν να επαναλάβω Και πραγματικά ευχαριστούμε όσους εργάστηκαν για τους φακέλους αυτούς και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από συγκεκριμένες ερωτήσεις που μου απευθύνθηκαν. Παρόλο που δεν σχετίζονται όλες οι ερωτήσεις με το μηχανισμό αυτό σταθεροποίησης και με τις ρήτρες διασφάλισης. Μας ρωτήσατε τι, συμβαίνουν, ε, τι συμβαίνει με τον περιβαντολικό δικό χάρτη, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα όσα είχαμε ζητήσει από την Κολομβία και το Περού, το ψήφισμα του 2006 και όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία που αποδίδεται στον οδικό αυτό χάρτη εσείς στο Κοινοβούλιο. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι η Κολομβία έχει ήδη παρουσιάσει κάποια προκαταρτικά στοιχεία στον Μάριο Νταβίτ που είναι εισηγητής για την εμπορική συμφωνία και στον Μπέρντ Λάγκε για την ε, γνωμοδότης που συζητάμε τώρα και αποδεικνύει πως α, ε, τα παίρνουν αυτά όλα πολύ στα σοβαρά και ο πλήρης οδικός χάρτης μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμος. Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργό εξωτερικών θα συναντήσει τον κύριο Λάνκια για να συζητήσουν το θέμα. Δεν ξέρουμε ακριβώ τι συμβαίνει με το Περού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε συνεχή επαφή έτσι ώστε να υπογραμμίσουμε το πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια για μας. Και νομίζω πως και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε επαφή μέσω του εισηγητή σας με τη χώρα αυτή. Για το μηχανισμό σταθεροποίησης για την μπανάνα και για το κατά πόσο θα προστατεύσει τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, να πω τα Ξέρω πως οι περιοχές αυτές είναι εξαιρετικά ευάλωτες όταν έχουμε αύξηση απότομη των εισαγωγών. Και για το λόγο αυτό διαπραγματευτήκαμε τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά τους. Και ε, περιγράφουν και αντανακλούν την ε, πραγματική κατάσταση. Ακολουθούν ένα μοντέλο το οποίο έχουμε ε, χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, το οποίο έχουν βρει ικανοποιητικό και ελπίζω πως και εδώ θα ισχύσει το ίδιο. Αυτή η ειδική διασφάλιση θα ισχύσει και μετά τη μεταβατική περίοδο, δηλαδή αφού ε, διακοπεί η χρήση του ε, μηχανισμού σταθεροποίησης. Ακούσαμε και κάποιες ανησυχίες για το πώς θα τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Νομίζω ε, εκεί πια θα πρέπει να μας δώσετε ένα περιθώριο ευελιξίας. Μπορούμε να έχουμε υποκατάσταση, όπως είπε κάποιος. Αλλά εμείς τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά με ιδιαίτερη σοβαρότητα. τέτοια διασφάλιση δεν θα μπορούσαμε να τη δώσουμε μόνο στην μπανάνα για παράδειγμα, αλλά η Γαλλία μας έχει ζητήσει να παρακολουθούμε τις εξαγωγές ε, κορεατικών ε, αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό είναι κάτι αντίστοιχο. Όταν λοιπόν έχουμε παρακολούθηση τέτοιου είδους, και λαμβάνουμε έτοιμα παρακολούθησης, κάνουμε τις σχετικές έρευνες και μετά λαμβάνουμε μια απόφαση όταν ξέρουμε όλα τα στοιχεία του φάκελου. Το επαναλαμβάνω, μας ανησυχεί πολύ το θέμα αυτό. Εξετάζουμε ε, και το που βρίσκονται τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως πρέπει να δούμε και πώς θα καλύψουμε και τις ανάγκες ε, των απομακρυσμένων περιοχών. Θα το κάνουμε με ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση. Πρόσβαση στην, στα ταμεία προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να είμαι ειλικρινής για τις αντισταθμητικές αποζημιώσεις δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Τουλάχιστον για να αντισταθμιστεί η απώλεια σε μερίδια αγοράς στην περίπτωση αυτή. Για το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει εμεί μια πρόταση και εσεί ω συνομοθέτε θα αποφασίσετε. Εμεί εξετάσαμε τι θα συμβεί με την πλήρη απολευθέρωση ε, των εισαγωγικών δασμών ε, και αυτά πάντα στα πλαίσια των συμφωνιών του 2006 όπου η ποσόστοση αυξήθηκε ε, με τρόπο που ε, δεν θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να ε, επιδοτούμε ακόμα παραπάνω τους παραγωγούς μπανάν στις απομακρυμένες περιοχές Ευρώπης γιατί είναι η παραγωγή που λαμβάνουν τις μέγιστες επιδοτήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι πως για την ένταξη στα ΠΟΣΕΙ δώσαμε ε, αποζημίωση 279 εκατομμύρια το χρόνο, ευρώ το χρόνο για να εξαλείψουμε και τι αρνητικέ συνέπειε από τι εμπορικέ συμφωνίε με το Περού, την Κολομβία και την Κεντρική Αμερική. Νομίζω το ποσό είναι αρκετά σημαντικό. Θα συμφωνήσετε κι εσεί. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Για δύο λεπτά κατόπιν ο κύριος Λάγκε. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Επιτροπέ, τους επόμενους τέσσερις μήνες μας περιμένει πολλή δουλειά. Θέλουμε να διαμορφώσουμε έναν οδικό χάρτη για την ενίσχυση των συνθήκων εργασία, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών συνθήκων στις χώρες αυτές, αλλά να υπάρξει και ένα δίκτυο ασφαλείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω πως αυτά μπορούν να γίνουν, αλλά θα είναι δύσκολα. Οπότε σας παρακαλώ, κύριε Επιτροπέ, να στηρίξετε αυτό το έργο, εκεί όπου μπορείτε, ειδικά όσον αφορά τη συμμετοχή της κυβέρνησης του Περού. Έχω την αίσθηση πως εκεί πέρα το μήνυμα δεν το έχουν λάβει, δηλαδή το πόσο σοβαρά ε, τα εννοούμε αυτά τα οποία λέει το Κοινοβούλιο. Οπότε θα πρέπει να έχουμε έναν οδικό χάρτη από αυτές τις δύο χώρες και επίσης σας παρακαλώ να αναλάβετε έναν ενεργό ρόλο ενώπιον του Συμβουλίου για να καταλήξουμε σε μια εφαρμογή του κανονισμού αυτού σε κάποιο λογικό χρονικό διάστημα έτσι ώστε και τα δύο αυτά στοιχεία να είναι στη διάθεσή μας έτσι ώστε το Νοέμβριο να μπορέσουμε να τα ψηφίσουμε και τα δύο και επιτέλους να τελειώσει αυτή η υπόθεση προς το συμφέρον και των Ευρωπαίων αλλά και των ανθρώπων στην Κολομβία και το Περού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Επόμενο ομιλητή για δύο λεπτά, ο εισηγητή, ο κύριο Λάιχτφριντ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κράτησε λίγο καιρό αυτή η δουλειά και θα ήθελα τα δύο λεπτά αυτά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την καλή μας συνεργασία για τις συζητήσεις που είχαμε να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της γραμματείας για τη στήριξή τους και τους δικούς μου συνεργάτες στο γραφείο μου που ήταν υπεύθυνοι για αυτό το θέμα. Αρχίως νομίζω πως τα είπαμε όλα τα υπόλοιπα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ε, ήταν παρόντες για την παρουσία ε, τους και την συμμετοχή τους, τους διερμηνείς, ε, την γραμματεία. Καλή νύχτα σε όλους, η συνεδρίαση διακόπτεται. Η ψηφοφορία είναι αύριο στις 12 η ώρα. Καλή σας νύχτα.